Ήρθε η ώρα των ψηφοφοριών. Το, πρώτο σημείο είναι η σύσταση για δεύτερη ανάγνωση όσον αφορά τη θέση του Συμβουλίου σαν αυτά τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έκθεση της κυρία Γκορστέτ και θα ψηφίσουμε τη θέση του Συμβουλίου. Λοιπόν, πρώτο, πρώτη ομάδα τροπολογιών υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε η θέση του Συμβουλίου θεωρείται ως εγκεκριμένη και ως τροποποίηθη. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Γκροστέτ. Το επόμενο θέμα είναι η πρόταση ψηφίσματος που αφορούσε τις ε, θελοντικές συμφωνίες συνεργασίας όσον αφορά το νόμο για τα δάση, τροπολογία 3, 1, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχές έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να γίνει και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Τροπολογία 3. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Απερίφθη. Ψηφίζουμε την πρόταση ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Ζαντό με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον εισηγήτη μας. Δεύτερη έκθεση του κυρίου Ζαντό. Ξανά ονομαστική ψηφοφορία. Μάλλον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια ξανά στον εισηγητή. Επόμενο θέμα. Πρόταση ψηφίσματος για τις εταιρικές συμφωνίες με τις χώρες του ειρηνικού. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεν είναι καθαρό το αποτέλεσμα. Ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος την τροπολογία 5. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση ψηφίσματος ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. έκθεση του κυρίου Μάρτιν όσον αφορά την προσωρινή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του Ειρηνικού. Έχουμε σχέδιο ψηφίσματος, δεν υπάρχουν τροπολογίες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον κύριο Μάρτιν. Επόμενο θέμα. Ψηφίζουμε πέντε προτάσεις ψηφίσματος για διεθνή υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε την κοινό πρόταση ψηφίσματο στο σύνολό τη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όλες οι άλλες καταπίπτουν. Επόμενο θέμα, πρόταση ψηφίσματος για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Σερβίας. Τροπολογία 4. Έχουμε προφορική τροπολογία. Κυρία τσεκ. Θα ήθελα να υποβάλω προφορική τροπολογία στον αφορά τροπολογία 4 του Φρανσίσκο Μπραντ και εμένα. Το τελευταίο το κομμάτι θα το διαγράψουμε και πούμε καλούμε τη Σερβία να έρθει σε διάλογο με το Κωσυφοπαίδιο χωρίς να αναφέρεται σε διαπραγματεύσεις όσον αφορά το καθεστώς του Κωσυφοπαίδιο. Και ελπίζω να το υποστηρίζετε αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Φαίνεται να... Ο κύριος Πόσολτ. Θα ήθελα μόνο να συστήσω υπό αυτούς τους όρους να υπερψηφίσουμε. Thank you very much for that. Σας ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 4 ως ετροποποίηθη με ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 8 κατά, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα θα κάνουμε έλεγχο αν θέλετε. Λοιπόν, ας κάνουμε έλεγχο για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 8. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 11 έχουμε δύο τροπολογίες. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, θα γίνει έλεγχος. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, τροπολογία 5. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 6 έχει αποσυρθεί. Μετά την παράγραφο 12, τροπολογία 8, έχουμε προφορική τροποποίηση του κύριου Κατσίν. Κυρία Αντιπρόεδρε, Αντιάννα Βουάλη, λαμβάνοντα υπόψη τη σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα ήθελα να ονομαστική ψηφοφορία όσον αφορά την τροπολογία 8. Λόγω τη ατυχού αποφάσεω σερβική κυβερνήσεω, να μην παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο. Και απόφαση τη Μεσολαβητή της Σερβίας ε, που ήθελε να παραστεί υπέρ του σερβικού λαού. Είναι μήνυμα προς τη Σερβία και όλα ε, τα υποψήφια κάτι μέλη ότι δεν γίνεται παζάρα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να υπάρχει ευρεία υποστήριξη για αυτή την τροπολογία θέλω να υποβάλω και πολύ σύντομη προφορική συμβαστική τροπολογία που αρχικά είχε προετοιμαστεί από την κυρία Μαριαλένα Κοπά να πούμε το εξής λυπάται για την αρχική απόφαση της κυβερνήσεως να μην παραστεί στην τελετή απονομής του βραβείου Ειρήνης ε, Νόμπελ στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου. Καλωσορίζει όμως την πρωτοβουλία του Δημοσιολαβητή να παραστεί στην τελετή σαν υπεύθυνη και αξιέπαινη απόφαση. Παροτρύνω όλους τους συναδέλφους να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κατσίν. Θα ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα με την προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ε, αντιρρήσει. σε σχέση με αυτή την προφορική τροπολογία για να μπορούμε εδώ πέρα να εισαγάγουμε τη λέξη αρχικός, αρχική. Οπότε φαίνεται όχι. Okay, in that case the Ωραία, δεν γίνεται αυτό για την προφορική τροπολογία και τώρα όσον την ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει κάποια ένσταση για να διεξαγάγουμε ονομαστική ψηφοφορία. Είναι η δικαιωτική ευκαιρία δική μου το να την διεξαγάγω ή όχι. Για την τροπολογία 8. Ψηφίζουμε τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη κύριε Σφόποντα. Ναι, αλλά ψηφίσαμε την οκτώ, στην ονομαστική. Νόμιζα ότι μόνο την ονομαστική. Α. Amendment 1, those in favor. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπή είναι υπέρ, υπή είναι κατά αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος ή στο σύνολό του με ονομαστική ψηφοφορία τώρα. You voted. vote is now closed. Πέρας. And that is adopted. Εγκρίνεται. Και τώρα η έκθεση του κυρίου Κάτσιν όσον αφορά την ε, Συμφωνία είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωσης Σερβίας με μια ψηφοφορία ενιαία για όλο υπέρ κατά και αποχές. Και εγκρίνεται με ευρεία πλειοψηφία η συνεδρία κύριε Κάτσιν. Το επόμενο είναι η ψήφιση της εκθέσεως Μαρίσα Ματίας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την όσο του Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας. The vote, the vote is now open. Ψηφίζουμε. Body voted. The vote is now closed. Πέρασε. And that is adopted. Congratulations. Εγκρίνεται συγχαρητήρια, κυρία Ματίας. Το επόμενο. Πρόταση ψηφίσματος της ε, ε, Τρόπης Αναφοράς αφορά τους, τους εισπνευστήρες και τους αστηματικούς. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Next item is the vote on six motions for resolution on the situation in Haiti. One... Η κατάσταση στην Αϊτή, ένα χρόνο το σεισμό. Για το επόμενο ψήφισμα και θα το ψηφίσουμε τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το επόμενο θέμα είναι η ψήφιση του ψηφίσματος για παραβίαση εκ, ε, ελευθερίας έκφρασης και διακρίσεις ε, επί τη βάση προσανατολισμού σεξουαλικού στη Λουθουανία. Το έχουμε πρώτα την ε, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος υπαριθμών 2 σε δύο τμήματα, χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές. Για να κάνουμε έλεγχο τη για το δεύτερο ήμιση, ψηφίζουμε όσον αφορά τη δεύτερη παράγραφο, δεύτερο τμήμα αυτής. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραγραφός 5. Κατά διαίρεση είναι το πρώτο. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα, οπότε θα πρέπει να κάνουμε έλεγχο με ηλεκτρονική ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα του 5. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτωται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 5. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ, ψηφίστε. Όλοι ψηφίσατε πέρα. Απορρίπτεται. Και τώρα αιτιολογική παράγραφος α, υπέρ, κατά, αποχές α, και εδώ είναι οριακό το αποτέλεσμα οπότε θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. The Συγγνώμη, το 8, πρόκειται για το 8, όχι το α, 8. And Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, απόχέ. Γκρίνεται. Το λέγει παράγραφο παράγραφος σιγματάφ. Εύστρα λατινικά. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Και δόρυα το αποτέλεσμα μόνο στο πλέον ηλεκτρονικό έλεγχο όσον αφορά την τροπολογική. F ή σιγματάφ. Εψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Πέρασε. Και τώρα η αιτιολογική H ή ΙΤΑ, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Recital H, a check. If you open the Για το H ΙΤΑ θα γίνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Εψηφίσατε. Πέρασε. And that is adopted. So, the motion for resolution as a whole... Και τώρα το σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. And now the explanation. Και τώρα οι δηλώσεις, επεξηγήσεις της ψήφου.